So, bevor ich mich hier noch vergaloppiere, äh, in weiteren Ankündigungen Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Έγκριση ημερής διάταξης, ημερησίες διάταξης. Αναβάλλετε το σημείο 11, σας το λέω από τώρα. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς κυρία Αντωνέσκου. βάλετε το σημείο 11. Ωραία, το είπαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός εσθονικά και μαλτέζικα. Ακούστε προσεκτικά τώρα παρακαλώ όλοι. Τη Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε ακρόαση για το δικαίωμα στο νερό. Είναι η πρεμιέρα, θα σας στείλουμε και ιδιαίτερη γραπτή πρόσκληση, 3 με 6,5 το απόγευμα. Ήδη, εκτός από τους συνήθεις που έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, έχουν ζητήσει, ήδη από τώρα έχουν εγγραφεί 274 επισκέπτες που θέλουν να συμμετάσχουν. Δηλαδή φαντάζεστε το πανηγύρι που θα γίνει. Ε, θα έχουμε πολλούς προσκεκλημένους, θα είναι στην ίδια αίθουσα και πολύ θα χαιρόμουν να θα μπορούσα να καλωσορίσω και πολλούς βουλευτές. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Καλά, δεν μπορώ να αναγκάσω κανένα να έρθει στη συνεδρίαση, αλλά θα χαιρόμουν πάρα πολύ, το τονίζω, εάν ήταν ε, γεμάτες εδώ οι γραμμές και τα έδρανα των βουλευτών. Τι άλλο έχω να σας πω. Έχουμε την έκθεση COP19 από τη Βαρσοβία ε, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Στα έγγραφα ξέρετε που θα το βρείτε και που θα το ανακαλέσετε. Αποφασίσαμε στους συντονιστές να στείλουμε αντιπροσωπεία στην επόμενη διάσκεψη COP, COP20, που προετοιμάζεται ήδη. Και κύριε Σπυρίλο, από τις 11 έχει ομάδα επισκεπτών και ο Πέτερ Λίζελ αλλά θα τα πούμε τότε. 10 με 11. Θα τους ε, καλωσορίσουμε όταν έρθουν. Επόμενη ανακοίνωση. Έκτη, παρακαλώ. Ομάδα εργασίας υγεία, σήμερα 12 Φεβρουαρίου, 12.30 με 14.45. έχουμε εργαστήριο στην αίθουσα Α1, Ε2 για ένα σύστημα ευρωπαϊκό ενημέρωσης για τον καρκίνο. Επόμενη ανακοίνωση. Είχαμε ε, τριμερείς διαλόγους, ο πρώτος ε, στις 10 Φεβρουαρίου, ο δεύτερος για τις 6 Μαρτίου, ε, για, την, για τα απόβλητα και για τα διζητικά χωροκατακτητικά είδη. Χτες έγινε η πρώτη συνάντηση για τον τριμερή διάλογο και στις Μαρτίου. Και το επόμενο θέμα της κυρίας Μακάβεν στις 23 Ιανουαρίου έγινε ο πρώτος τριμές διάλογος και σήμερα θα γίνει ο δεύτερος. Εμπορία εκπομπών ρήπων ε, για τις αερομεταφορές. Πέτερ Λίζε, συνεχίζεται αυτό το σύριαλ. 18 Φεβρουαρίου θα γίνει η πρώτη συνεδρία του τριμερούς διαλόγου. Αυτά ήταν οι ανακοινώσεις του Προέδρου όλες αυτές. Ερχόμαστε στο τρίτο θέμα, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 25-26 Σεπτεμβρίου, 16-17 Δεκεμβρίου και 9 Ιανουαρίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνουν τα πρακτικά και ερχόμαστε στην ηχοστάθμη, στο θόρυβο των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο εισηγητή δυστυχώ κολλείται σήμερα και απουσιάζει, αλλά η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη τον αντικαθιστά επαξίως. Είμαι Ο νέος ούσκι. Θα σας διαβάσω ό,τι έγραψε. Ε, έχει και γραμματικά λάθη, δεν φταίω εγώ. Δεν το έγραψα έτσι. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για την ηχοστάθμη των ε, οχημάτων ένα σχέδιο συστάσεων για τη δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να παρουσιαστεί για έγκριση από την Επιτροπή ΕΜΒΗ. Η επίσημη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 25η Φεβρουαρίου. Ο συμβιβασμός είναι αποτέλεσμα δύσκολων διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να σας συστήσω στα μέλη της Επιτροπής να υιοθετήσετε το κείμενο όσο έχει υποβληθεί. Και δεν έκανα και την προφορά, ε. Νομίζω καλά το διάβασα. Ευχαριστώ πολύ για την ανακοίνωση αυτή. Στις 20 Φεβρουαρίου, σε δεύτερη ανάγνωση, θα το δούμε προθεσμία 25 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι για την κατάσταση των και στις 19 και 20 Μαρτίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, ενώ στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Όπως ένα σωρό πάει τον Απρίλιο. Λοιπόν, η θέση του Συμβουλίου μας έχει αποσταλεί ή θα μας τη στείλουν στη δεύτερη ε, Σύνοδο Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 24 με 27 το μηνός. Αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την έκθεση πιανού του κυρίου Ούρουτσεφ. Σημείο 5. Τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιώτου στη Σύμβαση Πλαίσιο των ΗΠΑ για την αλλαγή του κλίματο. Α, και 6 μαζί για την Τόχα και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι και αυτή του κυρίου Ούρουτσεφ. 5 και 6. Για την κλιματική αλλαγή και την αποκοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων. Το λόγο έχει ο εισηγητή. Thank you, Ευχαριστώ. Η τροπολογία της Ντόχα ε, δημιουργεί τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων υπό το πρωτόκολλο του Κιώτο που ξεκινάει από το 2013 και τελειώνει το 2020. Με, υποχρεωτικ... με δέσμευση για την υποχρεωτική μείωση των εκπομπών των αερίων. Η διάσκεψη, κλιματική διάσκεψη της Ντόχα ε, προσάρμοσε δύο αποφάσεις για την τεχνική προσαρμογή των δεσμεύσεων που αφορούν την, ε, τον, υπολογισμό των ε, μειώσεων. Έχουμε δύο νομοθετήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα εμπορίας εκπομπών και η απόφαση για τον επιμερισμό της προσπάθειας με την καταγραφή και την τεχνική διαχείριση, τους κάνονες δηλαδή για αυτά τα θέματα. Έχουμε επίσης εθνικά μητρώα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Μητρό για τις εκπομπές, για την καταχώρηση δηλαδή, των εκπομπών και την καταγραφή τους. Και η εφαρμογή του πρωτοκόλου του Κιώτο μετά το 2012 απαιτεί ε, μια δέσμη κανόνων για την τεχνική εφαρμογή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και της Ιρλανδίας και να εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση με το σύστημα εμπορίας εκπομπών και την απόφαση για τον επιμερισμό των, της προσπάθειας. Δεν θα μπω σε αυτούς τους κάνονες σε λεπτομέρειες. Ε, στην πρόταση της Κομισιόν εξηγούνται. Θα πρέπει να καλύπτουν διάφορους τομείς η διαδικασία που αφορά τις συναλλαγές του Κιώτο, με τις μονάδες ε, Κιώτο, που αφορά ε, την ε, αγορά, την απόσυρση κτλ. Επίσης, τη μετάβαση από, τη δεύτερη, από την πρώτη σε δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων. Ο τρίτος τομέας είναι η δημιουργία και οι τροπολογίες το, του αποθεματικού πλεονασμάτου της προηγούμενης περίοδου, καθώς και η περίοδος δεσμεύσεων, καθώς και η καταγραφή των ε, ε, εσόδων από τις συναλλαγές. Και η πρώτη διεθνής μεταβίβαση μονάδων Κιώτο. Η πρόταση της Κομισιόν στην αιτιολογική της σκέψη, το αιτιολογικό τμήμα, έχει και λεπτομέρειες και εξηγεί γιατί αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να συνταχτούν και δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω. Υπάρχουν όμως διάφορες πτυχές που θα ήθελα να τονίσω. Καταρχάς, καταρχάς να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, οι αβεβαιότητες, ποιες προσαρμογές πρέπει να γίνουν. Ε, τα ποσά των κρατών μελών καθορίζονται στην πρόταση της Κομισιόν, στην απόφαση της Κομισιόν για την επικύρωση της ε, Συμφωνίας της Ντόχα και οποιασδήποτε αβεβαιότητες ή προσαρμογές στον ορισμό του κοινού ποσού θα επηρεάσει μόνο το καθορισμένο ποσό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι τα ποσά των κρατών μελών, τα οποία είναι δεδομένα. Το άλλο σημείο. Κάποιοι διεθνείς λογιστικοί κανόνες δεν έχουν προσαρμοστεί επίσημα ακόμα. Δηλαδή, κανόνες καταγραφής καλύτερα οι σχετικοί διεθνείς κανόνες που διέπουν την καταγραφή των εκπομπών και την πρόοδο προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων έχουν συμφωνηθεί επί της ουσίας στην ε, Βαρσοβία τον Νοέμβριο του 2013. Αλλά η επίσημη προσαρμογή αναμένεται να γίνει στη Λίμα το 2014, το Δεκέμβριο το συμπεφωνημένο τμήμα αυτών των διεθνών κανόνων θεωρήθηκε ότι το έχουν αποδεχτεί όλα τα μέρη. Έχει κλείσει με τις δεσμεύσεις ε, στο πρωτόκολλο του Κιώτο για τη δεύτερη περίοδο. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτών των κανόνων, αλλά οποιασδήποτε ουσιαστικές αλλαγές θα πρέπει να απεικονίζονται σε καταξιοδότηση πράξης που θα έχει το δικαίωμα να συντάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελειώνω για αυτόν τον κανονισμό με το συμπέρασμα ότι το πεδίο του προτινόμενου, της προτινόμενης αλλαγής του κανονισμού για το μηχανισμό παρακολούθησης και αναφοράς των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απεικονίζει πλήρως την ανάγκη να συντάσσουμε και να προσαρμόσουμε συνεπείς κανόνες, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Αυτά για την πρώτη έκθεση. I would propose to have the discussion and after that to go to the... Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το σημείο και μετά να μπούμε στη δεύτερη έκθεση. Perhaps, ε, Ίσως ε, να τα συνδυάσουμε το 5 και το 6, τα δύο σημεία της ημερησίας διάταξης. Εγώ έτσι το θεωρώ πιο λογικό. Έτσι μου πρότεινε. Okay, I'll continue with the second one. Uh, Συνεχίσω λοιπόν και με το δεύτερο σημείο. Όσον αφορά την ε, τροποποίηση του κανονισμού στην Τόχα, εδώ πρέπει να γίνουν δεκτές αυτές οι προτάσεις από τους εταίρους του Κιώτο και φυσικά θα αρχίσει να ισχύει, θα τεθεί σε ισχύ μετά από την ε, αποδοχή από τα τρία τέταρτα των εταίρων του Κιώτου της ε, πρότασης. Δηλαδή η κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την αποδοχή του πρωτοκόλλου του Κιώτου. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά καθορίζει τους όρους της κοινή υλοποίησης ε, αυτών των ποτάσεων από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισλανδία. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω κάποια σημεία σε αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου. Καταρχήν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ βασιζόμαστε στο πακέτο την ενέργεια του 2009, δηλαδή σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών και το σύστημα του επιμερισμού. Εδώ το 20% της μείωσης των εκπομπών ε, έχει αποφασιστεί μέχρι το 2020. Στόχοι για τα κράτη-μέλη. Οι δεσμεύσεις, υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη ε, σύμφωνα με αυτό το πακέτο του 2009 δεν αλλάζουν με αυτή την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Δεν υπάρχει δηλαδή τροποποίηση όσον αφορά τους στόχους. Τα επίπεδα των εκπομπών, όπως καθορίζονται για τα κράτη-μέλη, καθορίζονται από την απόφαση αυτή του Συμβουλίου, παράρτημα 1, εγγραφό 1, η πρόταση της Επιτροπής δεν θέτει απόλυτους αριθμούς όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθότι το ποσό αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με τα συνολικά ποσά για όλα τα κρατημέλη και την Ισλανδία και αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος ο οποίος συνδέεται με αυτήν την αβεβαιότητα όσον αφορά το σύνολο του ποσού, καθότι και το ποσό το οποίο έχει καθοριστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει ο κίνδυνος εδώ ακριβώς επειδή το συνολικό αυτό ποσό θα καθοριστεί μόνο εάν υπολογιστεί το συνολικό ποσό. Η έκθεση αυτή ουσιαστικά εξαρτάται βεβαίως και υπόκειται στις ε, τροποποίησεις και την αναθεώρηση από τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρώ επίσης ότι το σύστημα εκπομπών, ε, εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθορίζεται εδώ από μια σχετική ευελιξία των μηχανισμών του Κιώτο. Όσον αφορά λοιπόν την πρώτη περίοδο αναφοράς, θα πρέπει να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολλές πιθανότητες να μη συμμορφωθεί σε σχέση με αυτό το πρώτο, την πρώτη αναθεώρηση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Όσον αφορά τη συμμετοχή των ε, τρίτων χωρών στο σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καταρχήν είναι η περίπτωση της Ισλανδίας, η οποία συμμετέχει σε αυτό το σύστημα εμπορίας των εκπομπών, ιδιαίτερα για την δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, δηλαδή το 2020, δηλαδή 13-20, και εδώ βεβαίως χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία μεταξύ των ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας. Άλλες τρίτες χώρες και η πιθανή συμμετοχή τους στο σύστημα πορείας ε, εκπομπών, χώρες που δεν ανήκουν στο σύστημα αυτό δεσμεύσεων, θα πρέπει αυτό να συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας. Τέλος, κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει ειδικέ ε, διατάξεις, προβλέψεις όσον αφορά τις, την τεχνική εφαρμογή της, τεχνικές εφαρμοστικές διατάξεις δηλαδή δεν περιέχονται. Εδώ θεωρείται ως προϋπόθεση ότι η συμφωνία της ΔΟΧΑ του Δεκεμβρίου του 2020 θα πρέπει να ε, υλοποιηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη της συμφωνίας. Οι τεχνικοί κανόνες θα πρέπει βεβαίως να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροποποίηση αυτής της πρότασης βασίζεται στην ε, προϋπόθεση ότι τα κράτη που έχουν δεσμευθεί είναι υπεύθυνοι για να τηρήσουν τους ε, όρους για όλες αυτές τις ε, συναλλαγές σύμφωνα με τα εθνικά μητρώα. Όσον αφορά μεταφορές ε, στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, στο διεθνές σύστημα, οι οποίες προβλέπονται από τα μητρώα του πρωτοκόλλου του Κιώτο, Εδώ έχουμε βεβαίως και τον ε, μηχανισμό αυτό του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Όσον αφορά δηλαδή τους στόχους και την αύξηση του βιπέδου αυτών των στόχων, ο μηχανισμός ε, του πρωτοκόλλου του Κιώτο όσον αφορά δηλαδή το να τεθούν υψηλότερα όρια αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί από κοινού από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρει πουθενά ε, με ποια διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια αλλαγή, μια τέτοια τροποποίηση. Και βεβαίως αυτό θα αποφασιστεί εάν και εφόσον προκύψει μια τέτοια περίπτωση. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι όσον αφορά την τροποποίηση της του πρωτοκόλλου του Κιώθου καθώς και την κοινή υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα όσον αφορά την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσει τα επίπεδα των εκπομπών, να πάρει μια απόφαση σε αυτό το τομέα και φυσικά εμείς στηρίζουμε το σχέδιο αυτής της ε, πρότασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα αρχίσουμε με την ε, συζήτησή μας, οι σκιώδεις συζητητές καταρχήν. Vas Άιχερτ. And first uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την ε, εργασία σας. Σας ευχαριστώ και για τις επεξηγήσεις που δώσατε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι και εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πολύ σύντομα να υιοθετηθούν, να προσαρμοστούν αυτές οι προτάσεις. Είναι καθοριστικό για μας και σας ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία επεξεργαστήκατε μέχρι τώρα το θέμα. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω για τα δύο θέματα στον εισηγητή αλλά και μια ερώτηση στην Επιτροπή. Στον εισηγητή θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την ουσία, το περιεχόμενο, έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό. Η τροπολογία 5, κατά κάποιο τρόπο όμως, προκαθορίζεται μια συμφωνία η οποία θεωρεί ως δεδομένη την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε, αν θέλετε, αυτό που ονομάζουμε μία φούσκα. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος ότι εδώ πρέπει να το καθορίσουμε ήδη το επίπεδο αυτό, γιατί κατά κάποιο τρόπο κρίνουμε πολύ αυστηρά τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν δυσκολία με την συμφωνία αυτή. Ως προς την ουσία, ε, φυσικά και θα συμφωνήσουμε, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εδώ χρειάζεται να μπει αυτή η διευκρίνηση. Πρόκειται για ένα νομοθετικό περιεχομένου ε, κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απαραίτητο να μπει εδώ αυτή η διευκρίνηση. Γι' αυτό και προτείνω εδώ να αλλάξουμε λίγο τη σύνταξη της τροπολογίας 5. Έχω και μία ερώτηση προς την ε, Επιτροπή. Αναφερόμαστε εδώ βεβαίως στο πρωτόκολλο του Κιώτο και τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται να δείξουν περισσότερη φιλοδοξία, να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τους στόχους τους. Και αυτό το 20% που έχουμε θέσει, αν κοιτάξουμε βεβαίως το χαρτιπορίας όπως έχει καθοριστεί μέχρι το 2020 και όλες τις μέχρι τώρα μελέτες κόστος ωφέλης που έχουν γίνει, διαπιστώνουμε ότι αυτά μάλλον θα επιτευχθούν. Η, ερώτηση λοιπόν που θέλω να κάνω προς την Επιτροπή είναι πώς θα προχωρήσουμε. Χρειάζεται αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου. Θα ήθελα λίγο περισσότερες διευκρινήσεις. Θα ήθελα να μην είμαστε τόσο άκαμπτοι στον καθορισμό που θέτουμε των στόχων γιατί ενδεχομένως για το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ε, θέσει πιο φιλόδοξους στόχους για το 2020. Τι έχει να πει γι' αυτό η Επιτροπή, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Βεβαίως το πιο σημαντικό και επανέρχομαι εδώ στην ουσία είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία μας, γι' αυτό και θα συνεργαστούμε στενά με τον εισηγητή για να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Κρίτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον εισηγητή και να το συγχαρώ για το έργο του. Είναι σε πολύ σωστή γραμμή και θα ήθελα να τονίσω, όπως και άλλοι συνάδελφοι, την ανάγκη να εγκριθεί ε, γρήγορα η έκθεση αυτή σύντομα για να μπορέσει ε, να συνεχιστεί η διαδικασία παλήθευσης. Και θα καλούσα και το Συμβούλιο να επιταχύνει τις διαδικασίες. Η πληροφόρηση μέχρι τώρα τι λέει, ότι το Συμβούλιο ε, προτίθεται να αποφασίσει από αυτού τον Ιούνιο ή ακόμα αργότερα. Νομίζω δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε να εμφανούμε υπεύθυνοι ε, απέναντι στην ΚΟΠ ε, του Παρισιού και της γαλλικής κυβέρνησης που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να το φέρει σε αίσιο πέρας, θα πρέπει να επιταχύνουμε όσο μπορούμε τη διαδικασία. Και αυτό θα είναι απολύτως απαραίτητο. Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο που δώσαμε στις αναπτυσσόμενες χώρες εμείς. Ήταν και το βασικό και μεγάλο αίτημα τους ε, χρηματοδότηση και κοιότο. Αυτά τα δύο. Ε, ε, εμείς δεχτήκαμε να τους ε, παραχωρήσουμε το Κιώτο 2. Ε, τώρα το θέμα της χρηματοδότησης είναι των κρατών μελών. Δεν έχουμε όλοι την ίδια χρηματοδότηση. Θα πρέπει το συντομότερο λοιπόν να κυρώσουμε αυτό το Κιώτο 2. Είναι πάρα, πάρα πολύ επίγον και σημαντικό. Θα κάνουμε και τροπολογίες. Βεβαίως δεν θα θίξουμε τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή, αλλά κάποιες αιτιολογικές σκέψεις που θα επηρεάσουν την εφαρμογή και ε, θα ε, έχουν σημασία κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Κάλαναν. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, δεν συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει και θα στείλει ισχυρό μήνυμα για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κύρωση αυτής της συμφωνίας. Ξέρουμε όλοι τα στοιχεία. Με ή χωρίς την Ισλανδία είμαστε στο 11% εμείς των συνολικών ρήπων. Και ε, μετά συυθύνουσα για το μέλλον. Επίσης γνωρίζουμε ότι η δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων για το Κιώτο λόγω των ε, κρατών που φεύγουν, που εγκαταλείπουν μετά την πρώτη περίοδο και κάποιων άλλων χωρών που δεν ε, δέχονται να δεσμευτούν θα καλύψει μόνο το 14 με 15% του συνόλου των εκπομπών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει η διαδικασία αυτή. Απλώς θέλω να τονίσω ότι ε, δεν χάλασε και ο κόσμος α πούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να μειώσουν ε, τις εκπομπές βάσει του διεθνούς καθεστώτος και νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει αντιστοίχως να φροντίσουμε οι νόμοι μας να ε, συμμορφούνται και να λειτουργεί σωστά ε, το σύστημα που έχει συμφωνηθεί. Μπορώ λοιπόν να συμφωνήσω ότι έχει σημασία να εγγυηθούμε τη ταυτόχρονη κατάθεση όλων των μέσων κύρωσης. Στη Λίμα στα τέλη του έτους θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα και κάποιες ανησυχίες θα τεθούν αναγνωρίζουμε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κάποια ευελιξία στη δράση της, υπάρχει ε, σημαντικός κίνδυνος να ε, ερμηνεύσει τις εξουσίες της με ευρία έννοια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, εδώ εννοώ τις κατεξουδότηση πράξης. όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά βλέπουμε την τάση να χρησιμοποιούνται κατεξουδότηση πράξης σε θέματα σαν αυτό που είναι καθαρά πολιτικό. Και κάποια στοιχεία για τις ενδεχόμενες ε, μεταφορές και ε, ένα σαφές crossover ε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε ας πούμε στην τροπολογία 2 που προτείνει ο εισηγητής οποιαδήποτε ελλείμματα ή πλεονάσματα αδειών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να είναι σε κατεξουδότηση πράξης. Μα αυτά είναι δικαιώματα των κρατών μελών. Νομίζω υπάρχει πρόβλημα εδώ και θα κάνουμε και κάποιες τροπολογίες σχετικά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Λεφεύρ, Κάτι σας ρώτησε ο κύριος Εκχάουτ. Ε, uh, Ευχαριστώ. Καταρχήν, όσον αφορά τα σχόλια του εισηγητή, όπως είπε στην ε, εισαγωγή του, Μιλήσαμε για τον μηχανισμό φιλοδοξίας, ambition mechanism του πρωτοκόλλου του Κιώτου, ουσιαστικά για χώρες που επιθυμούν να καθορίσουν νέους στόχους. Αυτό δεν προϋποθέτει επίσημη τυπική κύρωση. Η εφαρμογή όσον αφορά αυτών των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση αυτό, διότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτή η εφαρμογή, η υλοποίηση. Και σε αυτό αναφέρθηκε και ο εισηγητής. Δηλαδή μπορούν ατομικά και ξεχωριστά τα κράτη-μέλη να καθορίσουν πιο φιλόδοξους στόχους και μπορούν αυτό να το κάνουν. Προβλέπεται εξάλλου στο παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιώτου αυτή η δυνατότητα. Και να αλλάξει εξάλλου και το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να υλοποιηθούν πιο νωρίς. Οι αλλαγές αυτές των στόχων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέσω μιας διαδικασίας και μιας αλλαγής από μέρους των αρχών των νομοθετικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αλλάξει δηλαδή ο, φιλόδοξος, ο στόχος, η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρειάζεται μια νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί από τις δύο νομοθετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όσον το συνολικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, πώς ε, ανακοινώνουμε, κοινοποιούμε αυτό στα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει ένας μηχανισμός. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται επίσημη κύρωση όσον αφορά την αλλαγή των ατομικών στόχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει εδώ ότι χρειάζεται κατά κάποιο τρόπο να γίνουν δεκτές ε, μέσω των διαπραγματευθών να γίνει δεκτή μια άδεια όσον αφορά την αλλαγή αυτών των στόχων. Και αυτό θα πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, από τις δύο νομοθετικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περάσουμε δύο δηλαδή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τέλος ο εισηγητής. να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και για τις κριτικές που άσκησαν αλλά και για τη στήριξή τους. Καταρχήν για την τροπολογία 5 θα ήθελα να πω ότι και εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Μπορούμε λοιπόν να προσαρμόσουμε λίγο το κείμενο εδώ. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την ε, υιοθέτηση. Όσον αφορά το επίπεδο των τωρινών διαπραγματεύσεων, πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία κύρωσης ε, από μέρους του Συμβουλίου επικρατεί μια αβεβαιότητα. Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία στο Συμβούλιο Αυτά. Για τις τροπολογίες η προθεσμία είναι και για το 5 και το 6 και για τα δύο σημεία είναι στις 17 Φεβρουαρίου στις 12. 6 Μαρτίου θα ψηφίσουμε και για τα δύο και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε και για τα δύο σημεία. Και τώρα περνάμε στο θέμα της στρατηγικής για τα υνοπνευματόδη. Η Ρωμάνα Γιόρδαν είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ενόπνευμα δεν είναι κάτι που με έχει απασχολήσει, μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στο παρελθόν, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και χάρηκα που ήμουν και εγώ μέλος της ομάδας που εκπώνησε το ψήφισμα και την ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να πω ότι εξεπλάγει πάρα πολύ όταν διάβασα ότι η Ευρώπη είναι κατεξοχή περιφέρεια όπου οι πολίτες πίνουν, καταναλώνουμε το περισσότερο ενόπνευμα στον κόσμο. Καλά, από μόνο το αυτό δεν είναι ανισχυτικό, αλλά αν διαβάσει κανείς τα στοιχεία που δίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι η κατανάλωση νοπνεύματος έχει και συνέπειες στην υγεία. Και αυτό ισχύει και για την υγεία των Ευρωπαίων. Το 2006 εκπονήσαμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική μεν, αλλά αυτή εξέπνευσε πριν από λίγο γιατί ήταν εξαετούς διάρκειας και είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι απέδωσε όλες. Είχε κάποια αποτελέσματα, τώρα θα πρέπει να ζηθούμε τι μέλη γενέστε. δεν έχουμε πρόγραμμα δράσης ή στρατηγική δεν ισχύει πια και ακριβώς επειδή έληξε η στρατηγική θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα πρόγραμμα δράσης να την εθαρρύνουμε, όχι απλώς να την παρακαλέσουμε, να την παροτρύνουμε το συντομότερο να μας καταθέσει αυτό το πρόγραμμα δράση το αργότερο το Σεπτέμβριο. Επίσης έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μια νέα στρατηγική. Για ποιο λόγο. Στην ευρωπαϊκή κοινωνία έχουν επέλθει πολλές αλλαγές. Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι τα της κρίσης. Αυτό τι σημαίνει ότι η κατανάλωση πνεύματος έχει αλλάξει, οι συνήθειές μας έχουν αλλάξει. Ο κόσμος καταναλώνει περισσότερο ενόπνευμα για να ξεφύγει από τα προβλήματά του και από την κρίση. Η κρίση πλήττει περισσότερο τους νέους ε, που είναι και πραγματικά η πιο ευάλωτη ομάδα όταν συζητούμε για αυτά τα θέματα. Ε, του αλκοόλ. Γι' αυτό χρειάζεται και είναι τόσο σημαντική η νέα στρατηγική και θα πρέπει να έρθει το συντομότερο. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις βλαβερές συνέπειες του ινοπνεύματος. θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα και όχι να κάνουμε κάποιες γενικές δηλώσεις με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα πρέπει να προλαμβάνουμε την υπερβολική κατανάλωση του ινοπνεύματος, ιδιαίτερα ε, μεταξύ των νέων. Δεν θα πρέπει να προσθέσουμε νέο γραφειοκρατικό φόρτο και πρέπει να σας πω ιδιαίτερα ειλικρινά ότι αμφιβάλλω ότι θα βοηθήσει μια ε, μεγαλύτερη ε, επισήμανση δεν είναι θέμα ετικέτα. Και τώρα αν αγοράσει μια φιάλη πνεύματο, βλέπει την ετικέτα να γράφεται ε, ο αλκοολικός ε, βαθμός. Δηλαδή το να είναι πιο αναλυτική ετικέτα δεν θα αποτρέψει κανέναν από την κατανάλωση αλκοόλ. Ε, θέλω να ακούσω και τα επιχειρήματά σας και τα σχόλια των συναδέλφων. Ε, δεν έχω πρόβλημα αλλά τα μέτρα που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανονικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη συνειδητοποίηση για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης. Δεν ξέρουν οι νέοι πόσο ε, σοβαρές μπορεί να είναι οι συνέπειες όταν ε, αποκτήσουν αυτή τη συνήθεια να πίνουν τακτικά. Και ως γονείς θα πρέπει να προσέξουμε ε, να καταρτήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια βάση δεδομένων πολύ καλή, πολύ ενημερωμένη που να αναλύεται συνεχώς και να μοιραζόμαστε ε, βέλτιστες πρακτικές μεταξύ κρατών μελών. Η κατανάλωση του υγειονοπνεύματος όμως έχει να κάνει και με την εκάστοτε νοοτροπία, κουλτούρα και τις συνήθειες ενός κράτους μέλους, ε, εξού και είναι σημαντική εδώ η επικουρικότητα. Θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να γάρουν αυτά που τους αναλογούν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τα κράτη-μέλη. Ο Κρις Ντέβις. Uh, Ευχαριστώ. Σκιώδης, ο σκιώδης εισηγητής της ομάδας μας είναι η Ρεμπέκα, Ρεμπέκα Τέιλορ, δεν μπορεί να είναι μαζί μας και υποστηρίζει αυτή την έκθεση. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια εκ μέρους της. Ε, συμφωνεί με τη Ρωμάνα Τζόρνταν και η ανησυχία για την κατανάλωση ε, υνοπνευματοδών ε, από, από εκατομμύρια Ευρωπαίους και της οικογένειάς τους είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να τα κράτη-μέλη και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να κάνουν κάτι και να γίνει και κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ε, καταπολεμήσουμε αυτή την δαπανηρή μανία. Φυσικά αυτοί που πουλάνε αλκοόλ θέλουν να βγάλουν κέρδος. Το σημείο αυτό του ψηφίσματος είναι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή της. Κάποια δικά μου σχόλια. Ε, είμαι στο Google εδώ, καθώς ε, εξελίσσεται η συζήτηση. Πόσοι πεθαίνουν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι αποτελέσματα. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο και 320.000 νέοι πεθαίνουν προώρα από το αλκοόλ κάθε χρόνο. 75.000 Αμερικανούς κάθε χρόνο και μειώνει την ζωή ε, κατά 30 χρόνια των ε, ανθρώπων. Αυτό μου φαίνεται υπερβολικό. Αυτά είναι οι πηχαίοι τίτλοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 7.000 ε, άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο προώρα. Ή γιατί έχουν πιει μέχρι θανάτου ένα Σάββατο βράδυ. και μερικές φορές θεωρούνται και υποτιμημένα αυτά τα νούμερα. αυτό είναι, έρχεται σε αντίθεση με το ότι μπορούμε να το βρούμε παντού το αλκοόλ. στα σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μαγαζί. Αν το δούμε λοιπόν σε τη διαστολή με την ε, κάναβη που απαγορεύεται ε, και που δεν σε σκοτώνει, ποτέ δεν έχει σκοτώσει, ε, σκεφτείτε ότι άμα καταναλώσει καταναλώσεις κάναβη μπορεί να πας και πέντε χρόνια φυλακή. Αυτό που πει η Ρωμάνα, ε, οι εθνικές παραδόσεις, οι συνήθειες κτλ. Ε, δέστε τις ε, διαφορές ανάμεσα στη Σουηδία και στην ε, Ολλανδία για την ε, κάναβη. Ε, τελείως διαφορετικές πολιτικές έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές καταστάσεις στις δύο χώρες. το θέμα τελικά είναι πώς θα δούμε αυτή την ιστορία. νομίζω ότι εδώ πρέπει να παίξει ρόλο η επικουρικότητα, τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν δράση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιοριστεί. Δεν έχει μεγάλο ρόλο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν να τόσο Είμαι πολύ ευτυχής που έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με το θέμα. Αυτό ξέρουμε πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι το ενόπνευμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο κοινωνικά αλλά και προβλήματα σοβαρά στην υγεία. Είναι πολύ συγκεκριμένη σήμερα η σχέση που υπάρχει μεταξύ κατανάλωσης ινοπνεύματος και καρκίνου. Το καρκίνο του μαστού, το καρκίνο του του εντέρου. Και η σχέση μεταξύ των περιπτώσεων καρκίνου που έχουν από άτομα που καταναλώνουν ε, νόπνευμα είναι εμφανής και η έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι και φυσικά τα προβλήματα στην υγεία είναι εμφανή και σε πολλούς άλλους τομείς, τα καρδιακά νοσήματα, στο σηκώτη και η δράση μας εδώ φυσικά θα πρέπει να ενταθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν κοινέ πλατφόρμες συζήτηση ε, των θεμάτων αυτών. Το θέμα βέβαια του καθορισμού της τιμής είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν και πολύ διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει εδώ να δούμε όλοι πώς ε, διοχετεύεται στην αγορά, ποιο είναι το μάρκετινγκ των υνοπνευματοδών ε, ποτών, αλλά και η σήμανση. Πολύ ακόμα σήμερα δεν συνειδητοποιούν ούτε πόσες θερμίδες καταναλώνουν πίνοντας υνοπνευματόδη ε, ποτά, ούτε τις επιπτώσεις στην υγεία. Και χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ ότι οι πολιτικές ομάδες ε, στηρίζουν τις προτάσεις αυτές και ελπίζω πραγματικά για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα να καταφέρουμε να είμαστε φιλόδοξοι προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα όμως να δω μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μετά ένα πρόγραμμα δράσης και να μην ε, επαφιέμαθα τόσο πολύ στην αυτορύθμιση όπως κάνατε μέχρι τότε γιατί δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που ε, περιμέναμε. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποτύχει. Ποιο είναι ο στόχο του προγράμματο δράση, Είναι η συνολική μείωση τη κατανάλωση συνοπνεύματο. Συνολική. Όχι απλώς να ελαχιστοποιήσουμε τις βλαβερέ συνέπειε μεταξύ ε, κάποιων υποομάδων του πληθυσμού όπως είναι οι νέοι, οι έγκυε γυναίκε, ακόμα και οι αλκοολικοί. Έχει αρνητικέ συνέπειες στο σύνολο του πληθυσμού. Όπως υπενήχθηκε και ο Chris Ντέιβις αλλά πρέπει να σου πω ότι και ε, η κάναβη συνδέεται με τον καρκίνο του πνεύμονα, άρα δεν είναι το παρόν, θα το πούμε άλλη στιγμή. Υπάρχει και οικονομικός αντίκτυπος. Εγώ είμαι πράσινος και συνήθως σκέφτομαι ότι ο Ριπένον πρέπει να πληρώνει. Υπάρχει μια σουηδική μελέτη που λέει ένα λίτρο ε, καθαρού υνοπνεύματος 100% κοστίζει 90 ε, ευρώ στην κοινωνία, 800 σουηδικές ε, κορώνες. Δηλαδή κανονικά αυτός θα πρέπει να είναι και ο φόρος που θα ε, πρέπει να επιβάλλεται. Είναι υπερβολικό σε σχέση με τα σημερινά πρότυπα, αλλά είναι περίεργο που ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφηκε στο δικαστήριο κατά της Σουηδίας γιατί έχει πολύ ε, χαμηλούς φόρους στο ζήθος σε σχέση με τους υψηλούς φόρους στο νίνο. Ε, ενώ για το συγκεκριμένο δεν κάνει τίποτα. Και από το 2007 στο Συμβούλιο τα πράγματα έχουν αποτελματωθεί. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αυξήσει την ελάχιστη φορολόγηση του ινοπνεύματος, αυτό που τουλάχιστον θα πρέπει να κάνουμε κατά την άποψή μου είναι να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε την ίδια λογική που έχει επιβάλει το δικαστήριο στην απόφαση για την εισαγωγή από το διαδίκτυο. Δηλαδή ε, θα πρέπει το κράτος μέλος να έχει το δικαίωμα να επιβάλλει το φόρο, δηλαδή χώρα ε, προορισμού. Όταν κάποιος αγοράζει από το διαδίκτυο κρασί ή νόπνευμα, ε, λέει το δικαστήριο ότι θα πρέπει να εισπράττει η νοπνευμα λεει το δικαστηριο οτι θα κατανάλωσης τη διαφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί να μην ισχύει λοιπόν ο ίδιος κανόνας όταν δεν το παραγγέλνεις από το διαδίκτυο, αλλά πηγαίνεις ε, στην ε, αλλοδαπή για να αγοράσεις μόνος σου. Εγώ ζω κοντά στα σύνορα ε, της Σουηδίας με τη Γερμανία και ο κόσμος πηγαίνει στη Γερμανία και αγοράζει μέχρι και 200 ε, κιλά αλκοόλ και όταν πας και ένα ζευγάρι μπορείς να φέρεις μέχρι 400 κιλά και έχουν για δύο χρόνια ενόπνευμα και είναι ήσυχοι στο σπίτι τους. Βέβαια η Βίρα δεν κρατάει δύο χρόνια οπότε καταναλώνεται νωρίτερα και από νέους. Διότι την πουλάνε. Όταν πηγαίνεις ε, σε καταστήματα ε, παραμεθόρια, κανονικά αγοράζεις κάποια προϊόντα που δεν υπάρχουν στη χώρα σου. Ενώ στη Γερμανία στα σύνορα τα μαγαζιά είναι γεμάτα με υνοπνευματόδη για να πηγαίνουν οι Σουηδοί να αγοράζουν που είναι πιο φτηνά. Ορίστε, μπορούμε να έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση τη πολιτική υγείας. Ε, να μην έχουμε τόσες τεράστιες ποσότητες συνοπνεύματος που ο μόνος σκοπός τους είναι να αποφύγουν την υψηλή φορολογία. Και ε, παντού τρέχουμε να κλείνουμε παραθυράκια στη φοροδιαφυγή και στη φοροαποφυγή. Αλλά στην πολιτική για το ενόπνευμα τι έχουμε κάνει μηδέν στο πηλίκον. Να το σκεφτούμε. Δεν έχει νόημα ο κόσμος να πηγαίνει και να φέρνει ε, ολόκληρες... Ε, ποσότητες φορτία, φορτηγών και μάλιστα ε, μπορεί να αγοράζει και σουηδικό ένα πρόβλημα. Δεν ανάγκη να πηγαίνει στη Γερμανία να παίρνει γερμανικό. Εγώ ε, πρωτοστάτησα στις διαπραγματεύσεις και χαίρομαι που ήρθα σε αίσιο Κάτι άλλο έχει να κάνει με τη διαφήμιση ε, για το ενόπνευμα. Θυμάστε ε, στην Ευρωπαϊκή Τηλεόραση χωρίς σύνορα ε, διαφήμιση για το ενόπνευμα επιτρέπεται μόνο το βράδυ στην τηλεόραση. Και πάλι η ε, Γαλλία και η Σουηδία έχουν πολύ ισχυρούς κανόνες. Υπάρχουν όμως κάποια βρετανικά κανάλια στην Νότια Βρετανία που εκπέμπουν μόνο προς τη Σουηδία, δεν έχουν αγγλικό κοινό ε, και τι μπορεί να γίνει ένα διάβημα της Ιουδικής κυβέρνησης στη Βρετανική και τα λοιπά για να το λύσουμε μεταξύ τους. Αλλά είναι πολύ βαριά σχεδόν αφόρητη η κατάσταση. Εκρεμεί στο δικαστήριο μια υπόθεση εδώ και μια διετία και πλέον και δεν συμβαίνει τίποτα. Ε, θα πρέπει να πλουστεύσουμε αυτή τη διαδικασία. Να υπάρχει λογική όταν εκπέμπεις ένα τηλεοπτικό σήμα προ μία και μόνη χώρα, θα πρέπει να ακολουθεί την νομοθεσία του κοινού, του καταναλωτή, βλέπε. Ε, βέβαια, Άλλο είναι να εκπέμπει σε μια χώρα και να περνάει λίγο σήμα από τα σύνορα και να σε βλέπουν οι γείτονε. Εδώ ε, ε, ε, απευθύνονται εκπομπέ καθαρά στη Σουηδία, στι σκανδιναβικέ χώρε. Μπορεί η Ευρώπη να μην συμφωνεί για την ελάχιστη φορολογία και του συντελεστέ ή για ορισμένε πολιτικέ υγεία που συνδέονται με το ενόπνευμα, αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε να μην υπονομεύουμε ο ένα τη δουλειά του άλλου για τι βραβερέ συνέπειε του αλκοόλ. Και πιστέψτε με, η Σουηδία στο 1700 ήταν από τις πιο φτωχές χώρες και πήραμε δρακόντια μέτρα ε, γιατί ο πληθυσμός μας ήταν συνέχεια μεθυσμένος 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα για να αντέξουν τα βάσανα που ζούσαν. Ε, στη συνέχεια μετατρέψαμε τη χώρα μας, ε, τη μετασχηματίσαμε μεταξύ άλλων και την κάναμε πολύ καλύτερη χώρα. Τώρα γιατί να ξεχάσουμε αυτόν τον αγώνα στην Ευρώπη και να τον απεμπολίσουμε. Το πρόβλημα του αλκοόλ δεν είναι παλιό. Σε όλες τις χώρες υπάρχει. Τα γνωρίζετε κι εσείς. Εγώ σας είπα τι γίνεται στη χώρα μου. Σήμερα σε πολλές χώρες βλέπουμε ότι οι νέοι βγαίνουν και γίνονται λιώμα. Ε, ξέρουμε και για τις έγκυες είναι κακό το αλκοόλ. Αλλά φαίνεται ότι επειδή είναι και τμήμα της καθημερινής μας ζωής, δεν το καταλαβαίνουμε. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τη λογική ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη, αναλαμβάνεις και το κόστος. Στα τρόφιμα δεν γράφουμε ε, ότι έχει ινόπνευμα μέσα. Γιατί? Ένα μικρό ποτήρι κρασί έχει τις ίδιες θερμίδες με ένα ε, αναψυκτικό αεριούχο. Ε, ε, μιλάω για τις θερμίδες τώρα και για την παχυσαρκία και τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου που αναφέρθηκε. Αυτά. Ε, ήθελα να τα πω όμως γιατί ήταν πολλά. Μα, τους ξέρουμε, τους καλύτερους συναδέλφους έρχονται αργά και μιλάνε και πολύ. Ε, συγγνώμη κιόλας. Η κυρία Γιανακουδάκη, παρακαλώ. Θα είμαι πιο ε, σύντομη. Είσαστε Σουηδός, έτσι δεν είναι. Ναι, την εθνικότητά σας θα το μάθω. Τα κράτη-μέλη, η βιομηχανία και η ΜΚΟ θέλουν να γίνουν κάτι, μια ευρεία, πλήρη στρατηγική. Και είναι καλό ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το ψήφισμα ε, και να συμφωνήσουν όλες ε, οι πολιτικές ομάδες, όλα τα πολιτικά κόμματα. Είναι αμφισβήτητο ότι υπάρχουν επιπτώσεις ε, από το αλκοόλ στην υγεία. Υπάρχουν κίνδυνοι όχι μόνο σε αυτούς που πίνουν υπερβολικά, αλλά μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Ε, Παραδείγματο χάρη όταν μπαίνει και οδηγεί και μετά οδηγεί. Η στρατηγική Ευρωπα... ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βοηθήσει τι εθνικέ κυβερνήσει ε, και τη δράση του, ώστε να μειώσουν την ε, ζημιά λόγω αλκοόλ στου ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη τη, είναι εκεί για να βοηθήσει τι εθνικέ στρατηγικέ. Οι πράσινοι είναι λίγο ανήσυχοι για την επιρροή που θα έχει το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία ε, για αυτών που πίνουν. Ε, καλό είναι να τους έχουμε μαζί μας σε αυτή την πορεία, σε αυτό το εγχείρημα, παρά να προσπαθήσουμε να τους αποκλείσουμε. Θέλω να δουλέψω μαζί μας και ελπίζω ε, η έκθεσή μας να γίνει ακριβώς γι' αυτό πιο δημιουργική, πιο ισχυρή αυτό το σχέδιο για όλα τα κράτη-μέλη ε, με βρίσκει λίγο διστακτική, γιατί νομίζω ότι εκεί ακριβώ έχουν τι αρμοδιότητέ του τα κράτη-μέλη, παραδείγματο χάρη σε επίπεδο αδειοδότηση. Δεν θέλω να υπάρχει μια ελάχιστη τιμή επίση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί τσακ με μια τιμή να λύσει το πρόβλημα, αλλά μέχρι στιγμή μα βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στο ψήφισμα και ελπίζω να δούμε από κοινού τι ε, τροπολογίε, να τι περάσουμε, να τι συμφωνήσουμε, να τι περάσουμε και να γίνει ακόμα καλύτερη έκθεση. Κύριε Άντερσεν. Χαιρετίζω αυτή την πρόταση που αφορά το ενόπνευμα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι εδώ θέλουμε όλοι αυστηρότερα μέτρα, ιδιαίτερα για τους ανήλικους. Από μέρους της Ιρλανδίας υπάρχει το θέμα αυτό στην επικαιρότητα και φυσικά το θέμα Αυτό είναι και πάρα πολύ παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα αυτό είναι μια μάστιγα στους νέους οι οποίοι πίνουν τεράστιες ποσότητες ε, αλκοόλ σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βλέπουμε κατόπιν ότι αναφέρουν στα κοινωνικά δίκτυα τι ήπιαν και πώς διασκέδασαν, αν μπορεί κανείς να ονομάσει αυτό το πράγμα διασκέδαση. Βλέπουμε ότι και στην Ιρλανδία και στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το φαινόμενο ε, πλήττει τους νέους. Δύο νέοι ε, πρόσφατα έχασαν τη ζωή τους από υπερβολική κατανάλωση ινοπνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτού του είδους η διασκέδαση, το binge drinking, δηλαδή η κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ινοπνεύματος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είχε σημαντικά, σημαντικές επιπτώσεις. Πολύ πρόσφατα είδαμε νέοι να μεταφέρονται με νοσοκομιακά μετά από τέτοιου είδους διασκέδαση. Το ενόπνευμα λοιπόν μπορεί πραγματικά να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία. Γνωρίζουμε σήμερα εξάλλου και το κόστος για τη δημόσια υγεία που προκαλεί αυτή η υπερβολική κατανάλωση υνοπνεύματος. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε τη στάση μας, την ενημέρωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ θετική η πρόταση και ότι πρέπει να δείξουμε περισσότερη αυστηρότητα προς το φαινόμενο αυτό. Πρόεδρος, σας ε, ενοχλούμε. Να, ε, το συγγνώμη. Ο κύριος Μπόσον. Κολέγιτσε, κολέγε. Ε, <laughs> here I am. <laughs> Εδώ είμαι. Θα ήθελα να εκφράσω και τη δική μου ικανοποίηση που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως. Η κατάχρηση είναι και αυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Έχει σοβαρές επιπτώσεις ε, στην υγεία. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη επιπτώσεις στο σηκώτη οι οποίες δεν είναι ίσες στους άντρες και στις γυναίκες. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι οι γυναίκες ε, αντέχουν λιγότερο το ενόπνευμα Βλέπουμε επίσης ότι πλήττει διαφορετικά τις κοινωνικές ομάδες. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υιοθετήσουμε μια πολιτική η οποία θα ισορροπεί την κατάσταση όσον αφορά τα πλήγματα που προκαλεί το ενόπνευμα στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. μια πολιτική καταπολέμησης της ε, υπερβολικής χρήσης του ινοπνεύματος, η οποία βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσει από την πρόληψη, από την καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση, μια κοινωνική πολιτική, πολιτική στον τομέα της δημόσιας υγείας που φυσικά θα πρέπει να κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών αλλά και όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες για να βελτιωθεί το κείμενο αυτού του ψηφίσματος. Χρειάζεται αλλαγή στην πολιτική μας. Αυτό το έγγραφο είχε προετοιμαστεί το 2006 πριν την οικονομική κρίση και πιστεύω ότι σήμερα με την οικονομική κρίση τα κοινωνικά προβλήματα αυξήθηκαν και φυσικά αυξήθηκε και η αρνητική επίπτωση του Ινοπνεύματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα εδώ να συμφωνήσω η κατάχρηση Ινοπνεύματος έχει εξαιρετικά δραματικές συνθήκες, καταστρέφονται ζωές, καταστρέφονται οικογένειες, επιπτώσεις οικονομικές. Όλα αυτά τα ανέφεραν οι συνάδελφοι πριν από μένα. Ο Κρίς Ντέιβις είπε κάτι στο οποίο δεν θα συμφωνήσω όσον αφορά την κάναβη όταν λέει ότι δεν έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή. Επίσης αυτό που είπε ο Σλίτερ που αναφέρθηκε στο ιατρικό κομμάτι. Δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που αναφέρατε από επιστημονικής απόψεως γιατί και η κάναβης μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Οπωσδήποτε πάντως ε, επιπτώσεις στην υγεία. Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι δεν είναι τόσο βλαβερή ουσία. Εν πάση περιπτώσει το θέμα μας εδώ είναι το ενόπνευμα. Είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας ε, του ΕΛΚ εχθές και ήταν προφανές από αυτά που άκουσα από τους συναδέλφους ότι το θέμα της επικουρικότητας είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί βεβαίως εδώ στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές διαφορετικές ε, συνήθειες και παραδόσεις για το θέμα του ινοπνεύματος. Δεν μπορούμε λοιπόν εδώ να μιλήσουμε για στρατηγική, για τα ινοπνευματόδη. Θα πρέπει ίσως να αλλάξει ο τίτλος εδώ. Στρατηγική για την κατάχρηση των ινοπνευματοδών ποτών. Θα αποφασίσουμε σε δύο εβδομάδες για τον νέο κανονισμό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δώσουμε την ε, ε, εντύπωση ότι αλλάζουμε τα πάντα, ότι θέλουμε να απαγορεύσουμε τελικά την χρήση του ινοπνεύματος. Δεν πρόκειται περί αυτού, διότι μία λογική κατανάλωση ε, πνεύματο, το είπε εξάλλου και η προηγούμενη ομιλήτρια. Βεβαίω έχει διαφορετικέ επιπτώσει στην υγεία των ανδρών και των γυναικών, αλλά ας πούμε πέντε ποτήρια την εβδομάδα δεν είναι κάτι που πλήττει, αντίθετα μπορεί να επιμικίνει την ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Η κατάχρηση είναι το πρόβλημα και αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε. Και βεβαίως αυτό με ε, με χρήση λογικών ε, πρακτικών και μεθόδων. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Ε, θα πρέπει να βρεθεί συμβιβασμός για κάποια από τα σημεία. Παραδείγματος χάρη είναι το θέμα της σήμανσης. Έχουμε τα ε, όμορφα μπουκάλια κρασί με τις ωραίες ετικέτες. Θα πρέπει να επισημανθεί το θέμα των θερμίδων. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Επίσης έχουμε και την πρόταση από την Γαλλία να αναφέρεται ο κίνδυνος για τις έγκυες γυναίκες. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που... Είναι μια πρόταση εξάλλου της Γαλλίας που η οποία έχει υιοθετηθεί στη Γερμανία. Ε, είναι κάτι που ίσως δεν αναφέρεται επαρκώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Σουίτσα, ευχαριστώ πολύ. Ε, καλωσορίζω και εγώ αυτό το ψήφισμα και συμφωνώ περίπου απολύτως με τους συγητές. Ξέρουμε ότι ε, το κάπνισμα τα ναρκωτικά και το ενόπνευμα είναι τα τρία μεγάλα δυνάμα μάστιγες ολόκληρες που απειλούν όχι μόνο οικογένειες αλλά κοινωνίες ολόκληρες και οικονομίες ολόκληρες. Ακούσαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η κατανάλωση αλκοόλ και από την κρίση έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο. Αν είναι σωστά αυτά τα στοιχεία που δηλώνουν ότι αφορά 60 χρόνια νοσήματα ε, και πάρα πολλά χρήματα κάθε χρόνο για την καταπολέμησή τους. Και η υπερβολική κατανάλωση ε, αφορά μέχρι και 9 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σε οικογένειες που πλήττονται από αλκοολισμό. Οπότε έχει έρθει η ώρα να δράσουμε. Θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει ε, το συντομότερο ένα πρόγραμμα δράσης και θα κάνουμε και τροπολογίες για να βελτιώσουμε το ψήφισμα. Γνωρίζετε όλοι ότι αυτό είναι θέμα των κρατών μελών και επίσης η κατανάλωση πνεύματο σε κάθε χώρα εξαρτάται από την εκάστοτε παράδοση και κουλτούρα. Ξέρουμε ότι έχουμε τρεις ζώνες, αν θέλετε, γεωγραφικές. Στο νότο της Ευρώπης ο κόσμος πίνει μπύρα, ε, κρασί περισσότερο, στην κεντρική Ευρώπη μπύρα και στη βόρεια Ευρώπη ε, πιο σκληρά ε, ποτά. Το πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά και να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη. Από την άλλη, μην νομίζουμε ότι μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα κεντρικά και να, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κληθούν να τα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Βεβαίως να αναθεωρηθεί η στρατηγική, δεν διαφωνώ, αλλά να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριο Σπυρίλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φανταστικό το ψήφισμα που συζητάμε. Αν χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για να μειώσουμε τη ζημιά στην υγεία λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, αυτό είναι. Η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το σχέδιο, γιατί όπως διαβάσαμε ε, το αλκοόλ προ... προκαλεί και αρρώστιες, όπως διαβάσαμε, και ψυχιατρικές ε, ασθένειες. Ε, θα πρέπει να κάνουμε ευρεία ενημέρωση του κοινού, κυρίως προς τους νέους, όπου μετά από υπερβολική κατανάλωση νοπνευματοδών, συχνά είναι θύματα τροχιών ατυχημάτων. Επίσης, ε, οι γυναίκες που είναι έγκυες όταν καταναλώνουν αλκοόλ έχουν πολύ, πολλά προβλήματα και επίση θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο αλκοόλ. Θα πρέπει μαζί με τα κράτη-μέλη να συνεργαστούμε, Ευρώπη και κράτη-μέλη, όπως είπε κάποιος συνάδελφος, γιατί η υπερβολική χρήση αλκοόλ είναι ε, μία μάστιγα κοινωνική για όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, να ξεκαθαρίσω ότι κατά την άποψή μου, το είπε η προλαλήσασα, το νέο σχέδιο δράση δεν θα πρέπει να έχει έναν απλώς απαγορευτικό χαρακτήρα. Απλώς να μας μαθαίνει, να μας διαπαιδαγωγεί ε, για την σωστή χρήση του αλκοόλ. Με μέτρο. Πολλές επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια ε, και γνωσμένη χρήση του αλκοόλ, αλκοολούχων ποτών, παραδείγματος χάρη του κόκκινου κρασιού, είναι θρεπτικά τρόφιμα ουσιαστικά μίας ισορροπημένης διατροφής. Και κολλάει, πάει μαζί με τη, μεσογειακή, τη λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν θα παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ, Καλχάνης Φλόρενς. Προφανώς ε, υπογραμμίζω όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανείς γύρω από το ενόπνευμα. Πολύ ωραία τα είπε ο Πέτερ Λίζε και με μεγάλη ακρίβεια και σε καμία περίπτωση δεν τα αμφισβητώ. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, μα πρέπει η Ευρώπη να τα ρυθμίζει όλα τώρα, τα πάντα. Μετά από όλη αυτή την ιστορία με το καπνό, πρέπει να βάλουμε τώρα με το κρασί. Για να πάμε να τα εξηγήσουμε στους πολίτες μας. Και θέλω να είμαι και παρόν από καμιά μεριά να σας βλέπω πώς θα τα εξηγείτε στους πολίτες. Τι μπορεί να κάνει καλύτερα η Ευρώπη από τη Ρώμη, το Ελσίνκι, το Βερολίνο ή οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα. Και να πω και κάτι άλλο. Ίσως επειδή είμαι εδώ ο πρεσβύτερος, δεν είμαι ε, ε, ηθικολόγος ή δεν θέλω να πω τίποτα κοπλαστικό, αλλά τώρα θα λέμε αυτό απαγορεύεται, το άλλο απαγορεύεται, οι γονείς. Ε, εγώ έχω τρία παιδιά ο ίδιος που εντάξει μπορεί να έχουν αδυναμίες αλλά δεν χρειάζεται να τρέχω από πίσω τους να τους τα εξηγώ όλα. Έχω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Τώρα να αναθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι. Δεν πρόκειται να την ξεφορτωθούμε ποτέ. Δεν ξέρω, εγώ έχω τεράστιες επιφυλάξεις. Και δεν θέλω να ε, αφαιρέσω την ευθύνη από τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ζέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σημαντικό σε αυτό το θέμα, μην τα βλέπουμε άσπρο-μαύρο. Είναι νόμιμο ναρκωτικό το ενόπνευμα. Και στην Ευρώπη κάθε χώρα μέλος έχει ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερες εμπειρίες, οι κοινωνίες μας έχουμε να μάθει να το αντιμετωπίζουν με τελείως διαφορετικές ε, ε, καταστάσεις. Ε, μας είπε στη Βόρεια Ευρώπη, κύριο Σλούτερ, τι γινόταν και ε, στο παρελθόν ε, που ήταν μεγάλη κατανάλωση και με ισχυρή φορολογία μειώθηκε, αλλά είναι διαφορετική κατάσταση στην Ιταλία, στην Ελλάδα ε, και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Συμφωνώ και με τον Καρλ Χάιντς Φλόρεντς. Δεν θα πρέπει τώρα να κάνουμε αυτό το σφάλμα. Μια στρατηγική για το ενόπνευμα ή μέτρα ολόκληρα για το ενόπνευμα. Πιστεύω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε μεν, και να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι εμπειρίες μας και πώς από κοινού ε, θα βγάλουμε κάποια διδάγματα. Και ιδιαίτερα την ε, υπερβολική κατανάλωση, την κατάχρηση ε, αλκοόλ. Κατάχρηση ορίζεται διαφορετικά στην Αγγλία, στην Αυστρία ή στην Σουηδία γιατί είναι τελικά διαφορετικές και οι συνθήκες και οι συνήθειες κατανάλωσης συνοπνεύματος, πόσο πίνει ο κόσμος. Στην Αγγλία βγαίνουν ε, το Σαββατοκύριακο και καταναλώνουν τεράστιες προσπα... Ε, ποσότητες αλκοόλ. Ε, σε άλλα μέρη είναι πιο ισόρροπη η κατανάλωση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ε, και η μέση όρη είναι πάρα πολύ παραπλανητική σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάχρηση, η οποία κατάχρηση ορίζεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και θα ήταν ένα στρατηγικό σφάλμα και παραμονή εκλογών τώρα τέτοια ε, ώρα, τέτοια λόγια. Πιάσατε το καπνό, τώρα θα σας πούνε πιάσατε και το ενόπνευμα. Είναι πολιτικό το στοιχείο αυτό και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πάρα πολύ. Ναι, να συμφωνούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την κατάχρηση σε ορισμένες ομάδες στόχους, τι κάνουμε με την νεολαία. Είναι πρόβλημα στη χώρα μου ότι πάρα πολλοί ε, νέα κορίτσια και αγόρια βγαίνουν το Σαββατοκύριακο και ε, πίνουν υπερβολικά. Το θέμα δεν είναι να απολαμβάνει το αλκοόλ, αλλά να, πέ, πιείς μέχρι να πέσεις λιπόθυμος. Ε, αυτό θέλει αντιμετώπιση. Ε, καλή είναι η ενημέρωση, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Τώρα όταν βγαίνει ένα κορίτσι 13 χρονών και πίνει μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο χρειάζεται να απαντήσει το κράτος. Ε, η νεολαία ναι. Το δεύτερο που αναφέρθηκε ήταν οι έγκυες γυναίκες, βεβαίως μπορεί να προκαλέσει αυτό βλάβες στο έμβριο. Θα πρέπει και εδώ να ενημερώνουμε τις γυναίκες και είναι υποχρεωμένος ο νομοθέτης. Η, η μεθυσμένη οδηγή. Υπάρχουν πολύ υψηλά πρόστιμα στην Αυστρία και θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Μηδενική ανοχή. Αυτό που δίδει στην Αυστρία. Και ένα τελευταίο. Ναι στη σήμανση με μερικές εξαιρέσεις εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να, να... δεν πρέπει να αναφέρεται η θρεπτική αξία, οι θερμίδες δηλαδή πάνω στη φιάλη. Ο κόσμος ξέρει τι τρώει και πίνει και ένα ποτήρι κρασί, μια φιάλη κρασί δεν ξέρω ή ένα ποτήρι μπύρα, αλλά δεν ξέρουν πολλές φορές πόσες θερμίδες έχει αυτό και θα πρέπει να ενημερώνονται. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη, αλλά και τα κράτη-μέλη να υποχρεούνται. Για μακροπρόθεσμα, αν τα κάνουμε αυτά, θα κάνουμε το σωστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κρίστιν Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω το κείμενο και όντως υπάρχει ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσουμε την στρατηγική μας Υπάρχει η ενιαία αγορά, υπάρχει η ενιαία αγορά εινοπνεύματος που όπως ξέρουμε κυκλοφορεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν μια κοινή αντιμετώπιση και ένας κοινός ορισμός, μια κοινή σήμανση όσον αφορά τα ενοπνευματώδη σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα των θερμίδων επίσης. Πόσες θερμίδες περιέχει ένα μπουκάλι κρασί. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και σε καμιά περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει περισσότερο ευρωσκεπτικισμό και από τη στιγμή που χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες μπορούμε να έχουμε την ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Ευχαριστώ. Από τον Μάριο Πυρίλο ήρθαν οι επισκέπτες του Μάριο Πυρίλο, μάλλον θα ήθελα να τους καλωσορίσω θερμά. Ja. Sie, Sie haben es, glaube ich, aufgesetzt. Gut. Wir kommen jetzt. Ωραία. Και τώρα να περάσουμε στην Επιτροπή. Ο κύριος Ζουρού. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Thank you, Mr. Chair. Uh, first, I... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή που υπέβαλε το κείμενο αυτό, το ψήφισμα αυτό. Πολλοί από τους ομιλητές αναφέρθηκαν στο τεράστιο πρόβλημα που προκαλεί το ενόπνευμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε πολύ λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την δημιουργία μιας κοινή πολιτικής στον τομέα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και για μένα να αναφερθώ στο ρόλο των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση της μέχρι τώρα στρατηγικής. Η στρατηγική λοιπόν αυτή καθεαυτή δημιούργησε μια επιτροπή Όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές ε, στον τομέα του ενοπνεύματος, εδώ και χρόνια λοιπόν τα κράτη-μέλη συζητούν τις πρακτικές τους, τις προτάσεις τους, τις παραδόσεις τους στους διάφορους τομείς που αναφερθήκατε στη συζήτηση αυτή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας για τον καθορισμό της μελλοντικής ε, στρατηγικής και πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το αναφέρω είναι ότι αυτή η Επιτροπή ασχολείται στα διάφορα σχέδια, σε διάφορα προγράμματα όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτό που αναφέρεται, το φαινόμενο που πλήττει τους νέους αυτής της υπερβολικής κατανάλωσης ε, ινοπνεύματος σε ένα συγκεκριμένο και πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το περίφημο binge drinking, και μια κοινή δράση των κρατών μελών είναι κάτι που φαίνεται σήμερα να έχει γίνει αποδεκτό από όλους, από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την προσπάθειά σας, για το ψήφισμα αυτό. Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή βάση για μας για τη συνέχιση της συζήτησης στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής που επεξεργάζεται τις Εθνικές Στρατηγικές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα για άλλη μια φορά και για δεύτερη φορά να χαιρετήσω θερμά τους επισκέπτες ε, του κ. Πυρέλο από την ε, εκλογική του περιφέρεια. Μπορείτε να ακούσετε αυτά που λέω στα Ιταλικά, ελπίζω. Ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Υπάρχει και η προφορική ερώτηση. Ποιος είναι υπέρ? Όχι ο Πίτερ Λίζε. Ναι. Κατά αποχές. Ωραία. Δεχόμαστε λοιπόν την προφορική ερώτηση. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 17η Φεβρουαρίου. Στις 6 Μαρτίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Απριλίου θα γίνει η τελική ψηφοφορία, όπως εξάλλου για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και τούμε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 8. Ο κύριος Σλίτερ έχει το λόγο. Uh, thank you also that we could bring this up today. We are many colleagues. Ευχαριστώ. Πολλοί είμαστε αμήχανοι με την απόφαση της Κομισιόν για κατεξιοδότηση πράξης. Που λέει, εντάξει ας επισημάνουμε τα πρόσθετα, αλλά μόνο για τα τρόφιμα. Όχι όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε άλλες μορφές. Αν κοιτάξουμε το ιστορικό της θέσης του Κοινοβουλίου για την επισήμαση, ε, στην ε, γενική ας πούμε, έκθεση του 2009, την έκθεσή μου, όλες οι πολιτικές ομάδες είπαν ναι, να το επισημάνουμε. Μετά είχαμε τα βιοκτώνα, τα ε, καλλιντικά. Αλλά δεν είπαμε ότι στα καλλιντικά, ας πούμε, ή μάλλον στα τρόφιμα. Δεν είπαμε ότι μόνο όταν έχει ένα νέο υλικό θα, θα επισημαίνεται. Όχι, για όλα είχαμε πει. Τώρα γι' αυτό λοιπόν έχουμε αντίρρηση. Γιατί όλοι είχαμε πει τότε ότι και αυτό είχε συμφωνηθεί με το Συμβούλιο. κανένα δεν είχε πει τότε ότι αν έχει ένα παλιό πρόσθετο ε, δεν χρειάζεται να το επισημάνεις. Όχι. Θεωρούσαμε ότι όλα όσα είναι παρόντα σε μορφή θα πρέπει να επισημένονται. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αντίρρηση. Ο άλλος λόγος, αν δείτε τη μελέτη, λέει όπου είναι δυνατόν πάνω από το 0,15%. Πριν από τρεις εβδομάδες ε, διάβασα ένα άρθρο ότι υπάρχουν, υπάρχει μια καλή μέθοδος για να ανοιχνεύσουμε τα ανανοηλικά, πιο ευαίσθητη από την ε, παλιότερη μέθοδο. Το να βάλουμε όμως το κατόφλι πάνω από το 50% είναι γελίο, είναι περίεργο. Ο σκοπός επισήμανσης δεν είναι να εντοπίσουμε τους κινδύνους. Είναι να ενημερώσουμε τον καταναλωτή. Όταν έχουμε προσθέσει νανοηλικά, νανοσωματίδια, επίτηδες, θα πρέπει να το ξέρει ο καταναλωτής, να το πεις. Γι' αυτό 50% είναι λάθος όριο, είναι υπερβολικά ψηλό. Αν βάζαμε 10% όπως είπε η Εύσα, τότε θα καλύψεις πολύ μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των προϊόντων. Είναι δύσκολο να τα μετρήσουμε. Κοστίζει να τα μετρήσουμε. Είναι αδύνατο να τα ελέγξουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι γιατί θα πρέπει να βάλουμε το κατόφλι στο 50%. Η απόφαση ανάμεσα στο 0,15 και 50 είναι τελικά πολιτική, όχι τεχνική ούτε οικονομική. Επομένως, το 10% όπως πρότεινε η ΕΦΣΑ, ίσως είναι ένας λογικός συμβιβασμός που όλα, και το κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δεχτούν. Εγώ θα ήθελα και χαμηλότερο, αλλά τουλάχιστον ένα 10% θα πιάσουμε την πλειοψηφία των υλικών που θέλουμε να καλύψουμε. Για αυτούς τους δύο λόγους έχουμε αυτή την αντίρρηση. Και δεν χρειάζεται να πω και τίποτα άλλο, γιατί ούτως ή άλλως μας υποστηρίζουν και πολλές ομάδες. Κύριε Φεντερικ Ρίς. Ε, euh, και εγώ συνυπογράφω αυτό το ψήφισμα των ε, φιλελεύθερων. Και πριν να μπω στο ψητό, δύο παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους ε, συμβούλους που ξανάβαλαν αυτό το σημαντικό θέμα επιτάπητος και μετά από την ε, μαζική ψηφοφορία μας την περασμένη ε, Πέμπτη στην Ολομέλεια για την ε, επισήμαση όλων των ειδών κρέατος, νομίζω ότι τελικά υπάρχει τρομερή διαφορά απόψεων ανάμεσα σε εμά και στην Κομισιόν. Γιατί πραγματικά αξίζει να υπάρχει διαφάνεια στην δικαιοθεσία. Το αξίζουν οι καταναλωτέ. Είναι σοβαρό το ψήφισμα, σοβαρά τα θέματα, δύο είναι τα πιο σημαντικά. Ε, θα πρέπει να σεβαστούμε τον νόμο για την ενημέρωση του καταναλωτή. Ε, δουλέψαμε πολύ όλοι μαζί για να το πετύχουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα πρόσθετα να υποφελούνται από παρεκκλήσει. Το εκτιμώντα G της επιλογική μας σχέση εξηγεί το γιατί. Η Κομισιόν με αυτή την παρέκκληση αποδυναμώνει τον νόμο από κάθε ουσία θα πρέπει να απαιτήσουμε αυτός ο κανόνας ετικετοθεσίας να επιβάλλεται και στα πρόσθετα. Γιατί ακούμε εδώ την βιομηχανία ε, και ακούμε την ε, Επιτροπή να γίνεται φερεφωνό ε, Υπάρχει μια γενική νεφελώδης κατάσταση για, την, για τη χρήση των ανοηλικών. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια για τα νανοηλικά στα τρόφιμα. Ε, όλα τα άλλα θέματα, η ενημέρωση του καταναλωτέ, ε, τα, καταναλω... τα καλλιντικά. Εγώ ήμουν εισηγήτρια σε μία από αυτά και θέλαμε, θέλαμε να ενημερώνουμε τον καταναλωτή. Γιατί να κάνουμε λοιπόν εδώ για τα τρόφιμα ένα βήμα προ τα πίσω. Και γιατί βάλατε αυτό το όριο στο 50% και όχι 10% φελπίν. τα οποία συστήνει και η ΕΦΣΑ. Δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κανένας τεχνικός λόγος, καμία τεχνική δυσκολία για να το κάνουμε. Ο, νομίζω ότι, ε, επομένως, εφόσον η απόφαση είναι πολιτική, εμείς έχουμε την... Είμαστε σωστοί, ε, εμείς είμαστε λογικοί. Κυρία Γκέρλινγκ, ε, δύσκολο ψήφισμα. Δύσκολο να φτάσουμε σε συμπεράσματα γιατί έχει διάφορα, α, διάφορους άξονες σκέψεις και επιχειρηματολογίες. Μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάποιο και να συμμεριζόμαστε κάποιον άξονα, αλλά όχι όλους. Η ομάδα μου ε, δεν το προσυπέγραψε. Ε, και δεν μας ρώτησαν κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων, θα προσβληθούμε. Όταν κοιτάω τα επιχειρήματα κάτω του 50% που υπάρχει και στον ορισμό της ε, Κομισιόν, νομίζω ότι δεν είναι πολύ τίμια η αναφορά στο γράμμα της ΕΦΣΑ προς την Κομισιόν ε, έγινε ε, μία πρόταση για 20% ε, για την ασφάλεια. Ε, δεν έγινε όμως στα πλαίσια της επισήμας των τροφίμων και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν ενημέρωση για τη χρήση των ανοηλικών, όχι για την ε, ασφάλεια ή για την καταλληλότητά τους. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη διάκριση να την έχουμε υπόψη μας. Δεν καταλαβαίνω ότι να εφαρμόσουμε ένα άλλο ε, κατόφλι και στο γενικό ορισμό των ανοηλικών θα προσθέσει κάποια επιπλέον ε, πληροφόρηση προς τους καταναλωτές. Επιπλέον μου είπαν, και φυσικά δεν ενημερωνόμαστε όλοι από τις ίδιες πηγές, εγώ όμως προσπαθώ να Ενημερώνουμε από διάφορες πηγές. Ε, ότι οι δοκιμές δεν μπορούν αξιόπιστα να προσδιορίσουν τα ποσοστά. Επειδή η ΕΦΣΑ λοιπόν λέει και μάλιστα λέει κάπου ότι ελήψη πληροφοριών συστήνουμε αυτό, νομίζω ότι αξίζει να το κάνεις μόνο αν το τεστάρεις και ξέρεις ότι αυτό είναι 10%, 20%, 30%. Αλλά δεν έχουμε τέτοια τεστ αυτή τη στιγμή, τέτοιες δοκιμές. Το να απαιτήσουμε λοιπόν επισήμανση από αυτή τη βάση θα ήταν προθύστερο νομίζω. Για το θέμα της πρότασης Κομισιόν να ε, ε, εξαιρέσουμε τα υπάρχοντα πρόσθετα στα τρόφιμα, θα έλεγα ότι για λόγους κοινή λογική πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κομισιόν. Καταλαβαίνω που το πάει, καταλαβαίνω τι λέει, εγώ ως καταναλωτή Αν κοιτάξω και εδώ το αγαπημένο μου πρωινό που τρώω εδώ και 10 χρόνια και ξαφνικά έχω ένα νέο ορισμό για τα συστατικά του, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στην σύσταση του, του, του, του δημητριακού αυτού, θα μου δημιουργηθούν περιττές ανησυχίες ως καταναλωτής. Καταλαβαίνω. και τη λογική αυτών που λένε, μα αυτό δεν λέει ο κανονισμός ε, για τα τρόφιμα. Αυτό λοιπόν το σημείο στο ψήφισμα θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Αλλά το υπόλοιπο δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Ε, γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχουν διαφορετικά πράγματα στο ψήφισμα, είμαι κατά γενικά του ψηφίσματος. Chris ναι, ευχαριστώ. Διαφωνώ με την κυρία Γκέρλινγκ, αλλά ε, θέλω να υπάρχει επισήμανση, αλλά το θέμα είναι τα κατόφλια ή τα ανώτατα όρια. Τι, είναι πρακτικό, ρεαλιστικό, ανοιχνεύσιμο στο κάτω-κάτω. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Πώς είπατε. Α, η κυρία Σαλτεμόζε. Α, δεν το κατάλαβα καλά. Πρώτα η κυρία Σαλτεμόζε, η Κρίστελ και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Όσα Βέσλοντ είναι αρμόδια από την ομάδα μας για αυτό το θέμα και απουσιάζει. Ήθελα από εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ότι υποστηρίζουμε το ψήφισμα και την αντίρρηση για τους λόγους που ανέφερε ο Καρλ Σλούτερ και θέλουμε να μάθουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επέλεξαν διαφορετικά όρια από εκείνα που προτείνει η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Πάντως υποστηρίζουμε την αντίρρηση και εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Äh, Ευχαριστώ. Ε, το Κοινοβούλιο. Ε, αν μου επιτρέπετε θα απαντήσω στα αγγλικά. Ε, σε ό,τι αφορά τα δύο σημεία τα οποία συνόψε ο κύριος Λούτερ ως βασικά στοιχεία του ψηφίσματος, που είναι η εξαίρεση ή ο αποκλεισμό ε, των προσθέτων και τα όρια, θα ήθελα να αποφασίσουμε το εξή. Και ως προς τις παρεκκλήσεις εξαιρέσεις που κάνουμε για διάφορα πρόσφατα, πρόσθετα, συγγνώμη, της κατεξουδότηση πράξης, κοιτάξτε, δεν είναι γενική απαγόρευση όλων των προσθέτων. Υπάρχει μια λίστα και δεν πρόκειται για όλα τα νέα πρόσθετα ή ε, όλες τις εγκεκριμένες ουσίες για να αλλάξει τελείως η παραγωγή ή η διαθεση οι διάφορες μέθοδοι. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό και να το τονίσω με ένα παράδειγμα. Ε, ο στιγμίος καφές. Από το 1946 περιέχει σιλικόνη συλλογικά, εν Η εξαίρεση έγινε για να μην υπάρχει σύγχυση στο μυαλό των καταναλωτών όταν βάλουμε τον όρο νάνο υλικά σε ορισμένα συστατικά και να νομίζουν οι καταναλωτές ότι ξαφνικά άλλαξε η σύνθεση του προϊόντος. Ενώ αυτό το προϊόν κυκλοφορεί από πάντα με την ίδια μορφή αυτή. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας επισήμανσης δεν θα μπορεί ο καταναλωτής να έχει μια επιλογή μετά λόγου γνώσεως, απλώς η σύγχυση θα οδηγηθεί. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού μεταξύ άλλων να υπάρχει ενημέρωση με νόημα για τους καταναλωτές και να μην παραπλανώνται. Για το όριο τώρα, το 50% συνάδει με ε, τον 696 κανονισμό του 2011 και τους αντίστοιχους ορισμούς. Το 2012 Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να μειωθεί αυτό κάτω από το 50% σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ε, εκτίμηση ασφαλείας των ανοηλικών. Σε ό,τι φορά λοιπόν τα όρια αυτά, Είμαστε σε πάρα πολύ στενή επαφή με το Κοινό Κέντρο Ερευνών και βασίσαμε το κείμενό μας ε, στις συμβουλές τους. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το όριο 10%. Αυτή τη στιγμή μπορεί να εφαρμοστεί. Και βάσει των συμβουλών και της ενημέρωσης που έχουμε λάβει από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, αυτή τη στιγμή ε, οποιοδήποτε κατόφλι κάτω του 50% δεν είναι εφαρμόσιμο γιατί δεν ανοιχνεύεται. Με τις μεθόδους που διατίθενται, τις αναλυτικές δηλαδή, αυτή τη στιγμή, νανοσωματίδια δεν μπορούν να μετρηθούν όταν είναι κάτω του 50% στα τρόφιμα. Αυτά μας λέγουν οι ειδικοί του κοινού ερευνητικού κέντρου. Όπως σας είπα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με χαμηλότερα κατόφλια ή ε, από το 50% στο 10%. Στην αιτιολογική σκέψη 13 της κατεσουσιοδότηση πράξης, το λέμε αυτό, ότι αν υπάρχουν ε, μέθοδοι στο μέλλον και εξελίξεις που θα επιτρέπουν να ανοιχνεύονται χαμηλότερες ποσότητες, να μειωθεί αυτό το όριο. Και επίσης δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε την ε, τοθεσία με την ασφάλεια του προϊόντος. Όποιον και να είναι το κατόφλι, 50%, 10% δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται να είναι εξασφαλισμένη ασφάλεια. Αυτό είναι έργο της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων και υπάρχει και σχετική νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα και για τα πρόσθετα στα τρόφιμα. Δεν θα αδειοδοτείται ένα προϊόν το οποίο δεν θα είναι ασφαλές. Ανεξαρτήτως ορίου. Συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι έχει κάνει υπέρβαση κατάχρηση εξουσίας με την κατεξουδότηση πράξη, ούτε η πράξη μειώνει την ε, ε, προστασία του καταναλωτού ή την ασφάλεια των τροφίμων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Davis. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Μας επιβεβαιώνει, μας λέει, ότι η προστασία των καταναλωτών διασφαλίζεται και ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί τίποτα κάτω από το 50% αυτό το όριο. Δεν ε, πιστεύω ότι μπορούμε εδώ να δεχτούμε την οποιαδήποτε νομοθεσία από τη στιγμή που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ότι δεν είναι εφαρμοστέα. Πώς μπορεί να απαντήσει αυτό η Επιτροπή. Ο Κάρλ Σλούτερ. να καταλαβαίνω τώρα τι λέτε όταν αναφερόσαστε στις εξαιρέσεις και λέτε ότι δεν καλύπτει τίποτα περισσότερο από αυτόν τον κατάλογο. Αυτό είναι ο κατάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ υλικό. Και μιλάτε για την αλλαγή μορφής. Παίρνετε το ε 171 ή το ε559 ή το 5-5-7. Οξύδιο μαγνησίου, σιλικόνης, οξύδια πυρητίου. Το θέμα είναι αν αυτά είναι παρόντα με μορφή νάνο υλικών και αν θα αυτό θα σημανθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πώς αυτό δεν έχει επιπτώσεις στην αγορά, στον ανταγωνισμό και αν αυτά υπήρχαν, προϋπήρχαν ε, στα προϊόντα ή όχι και ξαφνικά απλώς το αναφέρουμε στην σήμανση. Κάποια ναι, κάποια όχι. Ουσιαστικά αλλάζουμε τη σήμανση ενός προϊόντος ε, δεν καταλαβαίνω γιατί και δεν καταλαβαίνω τη λογική. Πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρεται αν η μορφή του είναι μορφή νανοηλικού ναι ή όχι. Μιλήσατε για το κατά πόσον αυτή η νομοθεσία είναι εφαρμοστέα. Πριν από τρεις εβδομάδες έμαθα ότι η μέθοδος έχει αλλάξει και ότι σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε τα νανοσωματίδια στα τρόφιμα. Ξέρουμε δηλαδή ποιο ποσοστό έχει μπει σαν πρόσθετα σε ένα τρόφιμο. Το θέμα είναι ότι Πώς μπορούμε να μετρήσουμε το προϊόν που αγοράζει κάποιος, πώς μπορεί οι μετρήσεις αυτές να ξέρουμε ότι είναι ε, ακριβείς, ότι τηρούνται αυτά τα ανώτατα όρια. Ναι, μπορεί λοιπόν να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία από τη στιγμή που μπορούμε να μετρήσουμε, να ανοιχνεύσουμε στα τελικά προϊόντα. Γιατί είναι λοιπόν αδύνατο να εφαρμοστεί το 10%, το 50%, όποιο και να είναι το ποσοστό, το πρόβλημα θα είναι το ίδιο. Το θέμα είναι ο καταναλωτής να μπορεί να έχει τις πληροφορίες που είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε. Δεν ε, έχω λοιπόν ε, θέμα εδώ, θέλω να μου εξηγήσετε αυτή τη λογική. Η Επιτροπή. Στο τελευταίο σημείο, αυτό που αναφέρατε για το όριο. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα. Το κοινό μας ερευνητικό κέντρο μας έχει βεβαιώσει ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει αξιόπιστη τεχνική μέθοδος όσον αφορά τη μέτρηση που αφορά αυτά τα νανοσωματίδια τα οποία θα, αν θέλετε, ξεπερνούν αυτό το 50% στο τελικό τρόφιμο, στο τελικό προϊόν. Αν δηλαδή κανείς θελήσει τελικά να διαπιστώσει ποια είναι η σύνθεση και ποια είναι η περιεκτικότητα σε αυτές τις ουσίες ε, ενός προϊόντος. Εγώ λοιπόν αναγκάζομαι σήμερα να βασιστώ στους τεχνικούς εμπειρογνώμονες, στο κοινό ερευνητικό κέντρο και λένε, επαναλαμβάνω, ότι κάτω από αυτό το 50% δεν μπορούν να έχουν αξιόπιστες μετρήσεις. και στη, σε μία από τις λέμε ότι αν δεν υπάρξει διαφορετική μέθοδος μέτρησης, δηλαδή νέα τεχνολογία, νέα τρόπος μέτρησης, θα παραμείνουμε σε αυτό. Όταν υπάρξουν νέα επιστημονικά δεδομένα, είμαστε διατεθειμένοι να ε, προσαρμοστούμε. Τώρα, το άλλο σημείο. Αναφερθήκατε σε αυτόν τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, κατοντάδες ε, πρόσθετα, αλλά όλα από αυτά δεν ε, εμφανίζονται με τη μορφή νανοηλικών και πιστεύω ότι και στο μέλλον αυτό δεν θα καλύψει όλα αυτά τα, ε, όλα αυτά τα πρόσθετα. Αναφερθήκατε στο οξύδιο μαγνησίου, πυρητίου. Πρόκειται για ουσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή επανεξετάζονται, επαναξιολογούνται από την ε, ε, Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΦΣΑ. Αν αυτή η επαναξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι η παρουσία ενός συγκεκριμένου μιας περιεκτικότητας, ενός ποσοστού νανοσωματιδίων αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, βεβαίως θα λάβουμε τα μέτρα μας. Με την σημερινή όμως κατάσταση, από τη στιγμή που υπάρχει η αξιολόγηση της ΕΦΣΑ όσον αφορά την ασφάλεια αυτών των ουσιών, εμείς θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί η αδειοδότηση. Όσον αφορά αυτήν τη συγκεκριμένη μορφή των ε, νανοσωματιδίων. Τώρα, εάν, εάν, εάν παραδείγματος χάρη για τα οξύδια πυρητίου Δύο συγγνώμη. Παρουσιαστεί με διαφορετική μορφή. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα θεωρηθεί σαν υπάρχον νανοηλικό, υπάρχον πρόσθετο. Αυτό το διοξίδιο πυρητίου θα θεωρηθεί νέο πρόσθετο, νέα ουσία, και σε καμία περίπτωση δεν θα μπει σε αυτήν την ε, κατηγορία εξαιρέσεων. Θα περιμένουμε την αξιολόγηση της ε, ΕΦΣΑ, της Υπηρεσίας Ασφαλής Οτροφίμων και θα είναι μια νέα κατηγορία, μια νέα σήμανση με ένα νέο αριθμό ε και σε αυτή την περίπτωση θα μπει η λέξη νάνο σε εισαγωγικά. Δεν πρόκειται για υπάρχον όμως νανό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση στα υπάρχον, στις υπάρχουσες ουσίες δεν θα χρειαστεί τέτοια σήμανση. Καλώς. Τελειώνει εδώ αυτή η συζήτηση και για την αντίρρηση θα ψηφίσουμε το απόγευμα στην ώρα των ψηφοφοριών. Ολοκληρώνει τη συζήτηση εδώ. Αν εγκριθεί σήμερα η αντίρρηση, στη δεύτερη σύνοδο του Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, εντάξει. στις 28 Ιανουαρίου ημερομηνία σας έχω στείλει ένα νέο επιστημονικό άρθρο που μπορούν σήμερα να μετρούν πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις από ό,τι στο παρελθόν με τη νέα μέθοδο. Αν δεν το έχει μάθει εύσα σας το λέω να το ξέρετε. Καλώς. Ολοκληρώθηκε είπαμε αυτή η συζήτηση. Και η μερίσια διάταξη για το πρωινό μας. Στις 3.30 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές μέχρι τις 5 και κλεισμένων των θυρών. Από τις 5 και μετά θα ψηφίσουμε την αντίρρηση πρώτα και άλλα θέματα. Καλό σας μεσημβρινό διάλειμμα.